Σύμφωνα με το άρθρο 105, τμήμα 6, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Προέδρων με ενημέρωσε, το πρόεδρο των Επιτροπών με ενημέρωσε ότι δεν έχει γύρει η αντίρρηση, η διάσκεψη πρόεδρων των Επιτροπών στη σύσταση της Επιτροπής ΕΝΒΗ να μην αντιταθεί στην εφαρμοστική πράξη. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μιας πολιτικής ομάδας ή ευρωβουλευτών στο κατώτατο τουλάχιστον όριο μέσα στις 24 ώρες, τότε η σύσταση θεωρείται εγκεκριμένη. Αλλιώς θα τεθεί στην ψηφοφορία. Η σύσταση υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Αυτή ήταν η ανακοίνωσή μου και περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης.